Αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις πριν δύο εβδομάδες, στη διάρκεια μιας συζήτησης στην Ολομέλεια, εκφράζαμε την ανησυχία μας όσον αφορά τη δραματική κατάσταση στη Συρία. Λίγες ώρες μακριά από το Στρασβούργο, οι Σύροι υποφέρουν, και είναι όμοιροι ενός παιχνιδιού